και διεθνείς συνθήκες που έχει ωστόσο κυρώσει η Λιθουανία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συζητήσει τα θέματα αυτά και να διασφαλίσει ότι αυτά τα πράγματα δεν θα συνεχιστούν. Ευχαριστούμε κύριε Ζιόπρο. Ολοκληρώσαμε τις παρεμβάσει διάρκεια ενό λεπτού. Και περνάμε στο τελευταίο σημείο τη ημερησία διάταξη. Παρουσίαση τη έκθεση Μποντή σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου. Κύριε Μποντής, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η έκθεση αυτή είναι καρπός της επικοδομητικής προσπάθειας που έκαναν οι διάφορες πολιτικές ομάδες. Προσωπικά τους ευχαριστώ τον κύριο Χάουλη, την, την κυρία Μπρέπολς και την κυρία Γιατενμάκη. Η έκθεση αφορά την σφαιρική στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσουμε στις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Συνεργασίας των Αραβικών Χωρών του Πευσικού Κόλπου. Η προσπάθειά μας ξεκίνησε εδώ και αρκετούς μήνες, πριν δηλαδή από τα τελευταία γεγονότα στον αραβικό κόσμο. Από τότε παρατηρήσαμε σε όλες τις χώρες της αραβικές τεράστιες διαδηλώσεις, οι οποίες διεκδικούν μεγαλύτερες, ε, περισσότερες ελευθερίες, περισσότερη δημοκρατία. Ήδη όμως πριν από την αρχή όλων αυτών των γεγονότων η έκθεση και οι τροπολογίες που είχαν γίνει δεκτές είχαν υπογραμμίσει όλα τα προβλήματα τα οποία προκαλούν αυτήν την εξέγερση. Έχουμε καταγγείλει όλες τις μορφές διακρίσεων και αυτές που βασίζονται στο φύλλο, στη θρησκεία Αναφερθήκαμε στο θέμα των εργασιακών δικαιωμάτων, των κοινωνικών δικαιωμάτων, την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία συνείδησης, τα δικαιώματα των γυναικών, την απαραίτητη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, την κατάργηση της θανατικής ποινής και των ακροτηριασμών και τον σεβασμό των πολιτικών δικαιωμάτων μπροστά στην καταστολή που ασκείται εις βάρος των διαδηλωτών και μετά από τη στρατιωτική μερικές φορές παρέμβαση των γειτονικών χωρών μελών του Συμβουλίου προετοιμάσαμε με τους σκιώδεις εισηγητές μία σειρά από προφορικές τροπολογίες οι οποίες στηρίζουν τους διαδηλωτές που πολεμούν για τη δημοκρατία υπογραμμίσαμε το θεμητό των διεκδικήσεών τους και καταγγείλαμε την βίαιη αντίδραση των καθεστώτων του Μπαχρέιν και την στρατιωτική παρέμβαση των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας που συμμετέχουν στις δυνάμεις καταστολής Εκφράζουμε λοιπόν τις βαθύτατες μας ανησυχίες απέναντι στην βίαιη αντίδραση του καθεστώτος και υποστηρίζουμε πλήρως την μεταβατική διαδικασία προς τη δημοκρατία. Είναι προφανές ότι η έκθεση αυτή καθορίζει και κάποιες μακροπρόθεσμες στρατηγικές προοπτικές αναφέρεται στις δυνατότητες μιας εταιρικής σχέσης με τις χώρες αυτές σε πολλούς τομείς γεωπολιτικούς, ενεργειακούς, εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς και περιφερειακής συνεργασίας. Και σε επίπεδο γεωπολιτικό το Ιράν είναι μια πραγματική απειλή ανάμεσα στο Ιράν και στο Ισραήλ οι χώρες του Περσικού κόλπου ε, σίγουρα θα είναι τα θύματα Μία τέτοια πιθανής σύγκρουση και περιμένουν από μας έτσι ώστε να αποτρέψουμε το Ιράν να αναπτύξει το πυρηνικό όπλο. Οι χώρες του κόλπου αντιπροσωπεύουν το 1 τέταρτο των μελών του Αραβικού Συνδέσμου και παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία και θυμίζω ότι είχαν προκαλέσει και την λεγόμενη Αραβική Πρωτοβουλία για Ειρήνευση. Σε επίπεδο ενεργειακό, το Συμβούλιο του Κόλπου είναι ο πρώτος παροχέας υδρογονανθράκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαρτώμεθα από τις χώρες αυτές, αλλά τα αποθέματα τους μειώνονται προετοιμάζουν την αλλαγή δραστηριότητας μέσω της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών και εδώ μπορούμε να τους προτείνουμε την εμπειρογνωμοσύνη μας σε εκπαιδευτικό και επιστημονικό επίπεδο οι χώρες αυτές θεωρούν ότι η εκπαίδευση είναι βασική τους προτεραιότητα. Υπάρχει έλλειψη πανεπιστημίων, έλλειψη διδασκόντων και ακριβώς βλέπουμε να εγκαθίστανται εκεί παραρτήματα των Αμερικανικών πανεπιστημίων. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ πίσω σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Σαν παράδειγμα μόνο 8 φοιτητές από τα, στις χώρες αυτές έχουν έλθει στην Ευρώπη τον προηγούμενο χρόνο στα πλαίσια του Έρασμος. Στα πλαίσια επίσης της περιφερειακής συνεργασίας το Συμβούλιο αυτό δεν προχωρά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με πολύ συγκεκριμένες εμπειρίες μπορεί να βοηθήσει να δώσει συμβουλές και εμπειρογνωμοσύνη. Και ζητάμε να υπάρξει και μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου που βρίσκεται σε επίπεδο επεξεργασίας εδώ και 20 χρόνια. Σας ευχαριστώ. Έχω δύο αιτήματα για ε, να λάβουν το λόγο δύο συνάδελφοι στην διαδικασία Catch the Eye. Ο πρώτος είναι ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ. Οι σχέσεις με το Συμβούλιο του Κόλπου έχουν μεγάλο δυναμικό και προσφέρουν πολλές δυνατότητες το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμούν να βελτιώσουν την συνεργασία. Εδώ είναι και το θέμα βέβαια της ικανότητάς μας να συνεργαστούμε με προσώπους των χωρών του ε, κόλπου περί προτεραιοτήτων και ταυτόχρονα να τίνουμε βίκο νου στα όσα έχουν να πούν. Σε πολλά θέματα έχουμε παρόμοιες απόψεις και γι' αυτό θα πρέπει η συνεργασία αυτή να μην περιοριστεί μονάχα σε εμπόριο και οικονομία. Όλοι γνωρίζουμε ότι η συνεργασία μας έχει ακόμα ανάγκη βελτιώσεων. Φιλόδοξες σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Συμβούλιο ε, Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου μπορεί να οδηγήσει και σε στενότερη συνεργασία και στενότερες σχέσεις με εκπροσώπους του μετριοπαθούς Ισλάμ στις σημερινές δύσκολες περιστάσεις αυτό θα σήμαινε ένα ακόμα πλονέκτημα της δραστηριότητας αυτής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πάσκα. Ο κύριος Σέγγεντη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ υποστηρίζω την ιδέα μιας ε, συμφωνίας συνεργασίας και ελεύθερων συναλλαγών με την με το ε, Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου που μπορεί να σημάνει σημαντικά πλεονεκτήματα λόγω των ε, αποθεμάτων πετρελαίου που διαθέτουν οι χώρες αυτές ε, υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, χρειαζόμαστε νέες εταιρικέ σχέσεις, νέους εταίρους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη παίζει σημαντικό ρόλο και ο σημαντικός αυτός ρόλος οφείλει να ενισχυθεί. Διαπραγματεύσεις γίνονται εδώ και έχουν αρχίσει εδώ και μία εικοσαετία. Πρέπει να ολοκληρωθούν επιτυχώς. Αυτό ωστόσο απαιτεί ευκαμψία, ευελιξία και από τις δύο πλευρές, διότι φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος αδιεξόδου. Χρειάζεται λοιπόν προσπάθεια αμφωτέρωθεν για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο και για να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταγωνιστική στο πλευρό των ΗΠΑ αλλά και της Κίνας. Χρειαζόμαστε σε ορισμένους οικονομικούς τομείς να βρούμε κάποιες ε, ειδικέ αγορές ώστε εκεί σε αυτές ε, να μπορέσουμε να αυξήσουμε το μερίδιό μας. Σας ευχαριστώ κύριε Σέγγετη. Η κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Μποντής για την έκθεσή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρετίζει την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων σε μια κρίσιμη φάση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες του κόλπου. Τα δεδομένα που προέρχονται από τον Μπαχρέιν δείχνουν ότι είναι απαραίτητο να εμβαθυνθεί η διεθνή συνεργασία. Οι έξι αυτές χώρες είναι ικανές να δείξουν ότι μπορούν να περάσουν σε μια ειρηνική μεταρρύθμιση της κοινωνίας τους με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η προμήθεια πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζεται από τα γεγονότα στις χώρες αυτές και γι' αυτό η συνεργασία ανάμεσα στην Ένωση και τις χώρες του Συμβουλίου είναι κάτι το απαραίτητο για να αποφύγουμε την αύξηση των τιμών σε διεθνές επίπεδο. Είναι πλέον καιρός οι 20 αυτοί ε, χρόνοι διαπραγμάτευσης να καταλήξουν ωφελώντα και τα δύο μέρη. Ο κύριος Επίτροπος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συζητούμε απόψε τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού ε, Κόλπου και από ό,τι ξέρω ζητήθηκε αναβολή για να, ε, επειδή υπάρχουν ε, σημαντικά, σημαντικές εξέλιξεις στον αραβικό κόσμο. Όταν ε, ξεκίνησε η σύνταξη ε, της έκθεσης, κανείς δεν ε, φανταζόταν πώς θα είναι σήμερα ο κόσμος, προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι των αραβικών χωρών και ολόκληρος ο κόσμος. Βέβαια, διαφέρει κάθε χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει την κάθε περίπτωση διαφορετικά, εξατομικευμένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να κάνει κρίσιμε επιλογές και να λάβει κρίσιμε αποφάσεις ε, είτε πρόκειται για τον Παχρέιν, τη Λιβύη, την Τινησία, ε, την Αίγυπτο κτλ. Κάποιες ε, υπάρχουν και, και διάφορες φιλοδοξίες και προσδοκίες και στο πολιτικο-οικονομικό επίπεδο. Υπάρχουν σημαντικά πακέτα. Πρέπει να να ανακουφιστεί ο, ο λαός ορισμένων από τον χώρο του Συμβουλίου Συνεργασίας από τα κοινωνικά προβλήματα. Πρέπει να γίνουν επίση εθνικοί διάλογοι με τη συμμετοχή όλων των πολιτών. Αυτά είναι κάποια θετικά που έχουν γίνει, αλλά έχουμε δει και κάποια βία επεισόδια. Στον Μπαχρέιν συγκεκριμένα. Παρακολουθούμε πρόσφατα ε, τα γεγονότα. Η Βαρόνια Άστον ε, πάρα πολλέ φορέ έχει εκφράσει την ανησυχία τη για την επανειλημμένη χρήση τη βία στου δρόμου. Υπάρχουν ε, μεγάλε τομακέ εντάσει. Επίση, πρέπει οι αστυνομικέ και άλλε δυνάμει που είναι επιτόπου να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα η Βαρόνια Άστον. Και πολλέ φορέ έχει ζητήσει να γίνει διάλογο, γιατί αυτό είναι ο μοναδικό τρόπο. Υπήρξαν κάποιες δημόσιες δηλώσεις, τις είδατε, υπήρξαν και άμεσες επαφές με Το θέμα τώρα για μας είναι πού οδηγούν όλα αυτά. Τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς πρέπει να ερμηνεύσουμε ε, τα γεγονότα. Είπε η κυρία Άστον ότι προτιμά τη δέσμευση αντί της ε, αδράνειας. Συμφωνώ. Ζητά περισσότερα έκθεση θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες ανταλλαγές και συναλλαγές μεταξύ επιχειρηματιών, για παράδειγμα. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να έχουμε πιο στενή επαφή και σχέσεις με τους ε, πολίτες των αραβικών χωρών και θα πρέπει επίσης να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε θετικά σε αιτήματα να διευκολύνουμε το διάλογο που θα οδηγήσει σε μεταρρυθμίσεις χωρίς αυτές δεν θα πρέπει να πάψουμε ε, να προασπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όχι όμως να επαγορεύουμε τα δικά μας ε, μοντέλα για τη δημοκρατία σε άλλες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει στεναρά ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να έρθουν από το εσωτερικό των χωρών αυτών και αυτό ισχύει και για τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού. Δεν θα πω εγώ στο Κοινοβούλιο τι θα κάνει σε σχέση με την έκθεση αυτή, αλλά πιστεύω ότι αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να το δούμε στρατηγικά το θέμα και ε, πρέπει να υπάρξει διάλογος. Αυτό είναι σημαντικό. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τη διαδικασία διαλόγου και μεταρρύθμισης. Να είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε στήριξη στις μεταρρυθμίσεις. Η ογνομοσύνη επίσης για την αντιμετώπιση ειδικότερων θεμάτων. Κάθε τέτοια δυνατότητα την επικροτούμε και τη χαιρετίζουμε, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν το ζητήσουν οι χώρε του κόλπου, αν ζητήσουν τη συνεργασία μα. Ε, μια λέξη για τη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών ε, με την περιοχή, που είμαι και άμεσα αρμόδιος γι' αυτό. Υπάρχουν κάποιες επαφές, θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα για να έχουμε εκπλήρωση των στόχων των εμπορικών ε, στο πλαίσιο και του Συμβουλίου Συνεργασίας. Βέβαια, η σταθερότητα φυσικά και είναι ένας, μια απαραίτητη προϋπόθεση και για να υπάρχει ο διάλογος, αλλά και για να υπάρχει μια ομαλή εμπορική ε, συναλλαγή. Σας ευχαριστώ και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μποντίσολος ιδιαίτερος. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, αύριο στι 11.30 θα ψηφίσουμε την έκθεση του κυρίου Μποντή. Έχω τώρα να ανακοινώσω στην Ολομέλεια ότι η Επιτροπή Οικονομικών και Νοσματικών Υποθέσεων μας ανακοίνωσε μία διόρθωση, διόρθωση κάποιων σφαλμάτων σε σχέση με το κείμενο το οποίο εγκρίθηκε στο Κοινοβούλιο. Η διόρθωση αυτή, το διορθωτικό, είναι στο Σιόνσον Direct, στην ιστοσελίδα αυτή. Θα συνεδριάσουμε εκ νέου την 5η 24 Μαρτίου, αύριο το πρωί 9 έως 1.